told me about that. Give him we have to talk about it. Colleagues, we now move to the declarations of vote. Den Stimmerklärungen, ich mache in der Muttersprache weiter im Interesse unserer Deutschen. Λοιπόν, θα μιλήσω γερμανικά. Η πρώτη έκθεση για την οποία θα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου, έκθεση Κινίτσι που αφορά ε, τις εγγύησεις ε, σχετικά με τα παιδιά. Η Κριστίνα Μόρβα για ένα λεπτό. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Ε, δεν ακόμη δυνατό να λάβουμε το λόγο. Ούτε εσείς ακούτε, γιατί μιλάτε με το διπλανό σας. Κανένας δεν ακούει. Νομίζω θα ήταν εξευτελισμός των Ευρωπαίων πολιτών να συνεχίσουμε τη συζήτηση υπό αυτές τις συνθήκες. Θα περιμένουμε να αποκατασταθεί η ησυχία και μετά θα μιλήσουμε. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να λάβουμε το λόγο. Πείτε τους ευρωβουλευτές να εγκαταλείψουν την αίθουσα της Ολομελίας αν θέλουν να έχουν ιδιωτικές συνομιλίες και να μην περάσουμε σε επεξηγής ψήφου αν δεν αποκατασταθούν αξιοπρεπείς συνθήκε για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Κυρία Μορβά, ήδη περίμενα μερικά λεπτά. Πάντως δίκιο έχετε. Θα κάνω αυτό που επισημάνατε. Παρακαλώ οι συνομιλίες να συνεχιστούν εκτός της αιθούσης, αγαπητοί συνάδελφοι. Κοιτάω και τους δικούς μου. Άνελη, Κάθριν, Σοφή, παρακαλώ. Οι συζητήσεις εκτός της για να μπορέσουν να εκφωνήσουν τις επεξηγείς ψήφους, ψήφου τους οι συνάδελφοι, παρακαλώ. I think that's So. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει τώρα. Κυρία Μορβάη, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ψήφισα υπέρ της έκθεσης Κινίτσι για τις δικονομικές εγγυήσεις των παιδιών που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Ίσως υπάρξουν κάποια προβλήματα με την ορολογία, γιατί με βάση τη συμβάση του ΟΗΕ, οποιοδήποτε κάτω των 18 θεωρείται ανήλικος. για μας ανήλικοι είναι 14-18, αλλά δεν εμπίπτουν στον ορισμό των παιδιών. Παιδιά για μας είναι κάτω των 14 και υπάρχει και αυτή η πιθανότητα να διώκονται δικαστικά. Αλλά πραγματικά όταν κατηγορούμε ένα παιδί, είναι ύποπτο ένα παιδί σε μια ποινική δίκη και επιπλέον δεν έχει τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε απροστάτευτα παιδιά σε τέτοιε ποινικέ διαδικασίε, γι' αυτό και υπερψήφισε την έκθεση. Ένα λεπτό, Γιουζι Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εγώ δεν υπερψήφισα την έκθεση για ένα βασικό λόγο. Ναι, μεν συμφωνώ ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια ενιαία προστασία των παιδιών σε ποινικέ διαδικασίε, αλλά δεν μου αρέσει και πολύ η οδηγία παρά είναι ευρύ το πεδίο εφαρμογής. Και μιλούμε και για την προστασία τη ιδιωτική σφαίρα. Αυτό όμω είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών κανονικά. Για παράδειγμα, στην Τσεχία, αυτή τη στιγμή συζητούμε το κατά πόσο παιδιά που διαπράττουν σοβαρά εγκλήματα θα πρέπει να κρατούν την ανωνυμία τους στις διαδικασίες. Επίσης, ε, το Κοινοβούλιο επέκτηνε τον ορισμό του ανηλίκου μέχρι τα 21 και σε αυτό εμπίπτουν και τα παιδιά. Γι' αυτό και δεν συμφωνούμε με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε κύριε Ποσπίση. Ο κύριος Μαμίκινς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κρίνοντας από τις ε, στατιστικές ε, πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε περίπου ένα εκατομμύριο παιδιά ε, μπλεγμένα σε ποινικέ υποθέσεις. Μεγάλος αριθμός ε, ύποπτων ή κατηγορούμενων παιδιών. Βέβαια τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα θέματα αυτά γιατί δεν έχουμε ενιαίο ορισμό για το τι εστί δίκαιη μεταχείριση του παιδιού. Η θέσπιση ελάχιστων δικονομικών εγγύσεων για τα παιδιά νομίζω ότι είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. Επίσης λέμε ότι η οδηγία εφαρμόζεται και για ανηλίκους ε, έως τα 21 έτη. Πιστεύω όμως ότι καλύτερα να διαβρύνουμε αυτήν την οδηγία ε, και να περάσουμε να εμπέσει το πεδίο εφαρμογή σε παιδιά από 14. Η συνάδελφο Γκίλντα παρετήθηκε από το λεπτό Πάμε στην άλφα Μακοβέη. Ευχαριστώ. Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά υφίστανται ε, διώξει μέσω ποινικών διαδικασιών, διώκονται ποινικά. Δηλαδή 12% του συνολικού αριθμού των υπόπτων ή κατηγορουμένων είναι παιδιά. Τεράστιος αριθμός. Επίσης, ε, οι δικονομικές εγγύησεις των παιδιών δεν εξασφαλίζονται. Ιδιαίτερα στις ποινικέ διαδικασίες και μάλιστα σε πολλά κράτη-μέλη. Παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Έτσι έχουμε διώξεις ε, ποινικέ παιδιών χωρίς να πληρούνται δικονομικές εγγύησεις από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ε, χρήσιμες λοιπόν είναι έστω και ελάχιστες ε, προδιαγραφές και δικονομικές εγγύσει για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Είμαστε υπέρ των δικονομικών εγγύσεων, υπέρ ε, του δικαιώματος σε δικηγόρο, σε νομική συνδρομή, δικαίωμα σε διερμηνέα αν χρειάζεται Γι' αυτό λοιπόν υπερψήφισε την έκθεση για να εξασφαλίζουμε δίκαιη δίκη και ελάχιστες κοινέ προδιαγραφές και δικονομικές εγγύησεις για παιδιά κάτω των 18 ετών που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενοι σε ποινικέ διαδικασίες. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Ντανιέλ Χάναν. Α, νάτος, κάτε μάλιστα και στη θέση μου. Έχετε το λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Η έκθεση αυτή βασίζεται στην χάρτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα, για θεμελιώδη δικαιώματα. Ένα έγγραφο το οποίο όταν το είχαμε διαπραγματευτεί, ο τότε πρωθυπουργό κ. Μπλερ είχε πει ότι δεν θα εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, μετά, ο σημερινός πρωθυπουργό είπε ότι ήταν σημαντικό να πάρουμε ένα ε, opt-out από την εφαρμογή του. Και πάλι τίποτα δεν άλλαξε. Βλέπουμε ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνουν τις εξουσίες στα χέρια τους. Παλιότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν διακυβερνητική οργάνωση για το εμπόριο και, την οικονομία. Ε, αλλά τώρα αποκτά η Ευρωπαϊκή Ένωση εξουσίες και αρμοδιότητες σε όλους τους τομείς. <laughs> Δεν μένουμε σταθεροί λοιπόν, ούτε καν στάσιμοι. Γι' αυτό λόγο πρέπει να φύγουμε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ομολογώ ότι δεν ψήφισα ναι, χωρίς δισταγμούς. Δεν θέλω η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει ευθύνε και αρμοδιότητε σε θέματα ποινικού δικαίου. Από την άλλη μεριά υπάρχουν ε, ωφέλη τα οποία υπερβαίνουν τα μειονεκτήματα, τις αδυναμίες και γι' αυτό το λόγο υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ότι ε, εγγυόμαστε η συμμεταχείριση για όλα τα παιδιά και τους δίνουμε δικονομικές ε, εγγυήσει έτσι ώστε να ε, μην ε, βρίσκονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια των ε, ε, ποινικών διαδικασιών. Και στην Τσεχία έχουμε ε, όρια για τα παιδιά που είναι παρόμοια αυτά που προτείνονται. Ευχαριστώ. Κέλλη, στηρίζω αυτή την πρόταση γιατί προστατεύει τα διώματα των παιδιών σε ποινικέ διαδικασίε. Εννιά συνεδρές του τριμερούς διαλόγου χρειάστηκαν ένα, ε, πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, είναι αντικείμενο τέτοιων διαδικασιών. Οπότε χρειάζονται εγγύησει για τα δικαιώματά τους. Πρέπει να προστατευθούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, να τους εξασφαλιστεί μια δίκαιη δίκη και κυρίως να αποφύγουμε ε, να ε, ξαναδιαπράξουν αδικήματα μέσω της κοινωνικής τους ένταξης. Σημαντική πρόκληση αυτό. Και πάλι καταδικάζω τις, ευρωπαϊκές, τις Αιγυπτιακές αρχές που, ε, ε, που ανέβαλαν την ε, δίκη του Μιλάλα, ο οποίος ε, είχε συλληφθεί πριν από τρία χρόνια ως παιδί και ακόμα δεν έχει δικαστεί. Ευχαριστώ. Ο Στίβεν Γουλφ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Πού και πού έχουμε ε, μία οδηγία που φαίνεται ότι έχει λογική διατύπωση ή φαίνεται και αποδεκτή. Και υπό, αυτές τις, ε, ε, υπό αυτούς τους όρους οι προτάσεις για δικονομικές εγγυήσεις για παιδιά σε ποινικέ διαδικασίες φαίνονται λογικές. το, Ευρωπαϊκό το Ηνωμένο Βασίλειο χειρίτερα αυτοεξαίρεσης για τη σχετική οδηγία, γιατί οι δικές μας ε, δικονομικές εγγύσεις είναι ψηλότερες για τα παιδιά από αυτές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν στις 23 Ιουνίου για το δημοψήφισμα ε, για την παραμονή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι σήμερα διαφορετικές οικονομικές διαδικασίες ε, για τα παιδιά υπάρχουν από τις δικές μας. Στην επαύριο θα έχουμε πάλι διαφορετικές από τις δικές μας νομοθετικές διατάξεις. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να υποταχθούμε και εμείς αυτούς τους κανόνες. Το θέμα δεν είναι το στάτου quo, το θέμα δεν είναι η παρούσα κατάσταση, αφορά το μέλλον. Και θα, αν παραμείνει το, Ευρωπαϊκό, το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνει σε κάτι που είναι απελπισμένο και σκοτεινό. Πάμε λοιπόν τώρα στην επόμενη έκθεση που αφορά στο σχέδιο προπολογισμού για το 2017. Πρώτος ομιλητή ε, για ένα λεπτό, ε, Λιγουάγα παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα ψηφίσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2017. Μας μένει ακόμη μια μακρά και χρονοβόρα διαδικασία για τη συγκρινοποίηση και γι' αυτό κρατήσαμε στάση αποχής για να παραμείνει ανοιχτό ο διάλογος πριν να κλειδώσουμε πλήρως τον προϋπολογισμό. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2017 δεν διδάχθηκε από τις εμπειρίες του παρελθόντος τίποτα. Θα έπρεπε να είχαμε πολύ πιο διωγγωμένο κοινοτικό προπολογισμό με έσοδα πολύ καλύτερα κατανεμημένα και που να στηρίζεται στο κατακεφαλήν εισόδημα των κρατών μελών πάνω απ' όλα. Τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την επιστροφή των προσφύγων και για, την, για το συνοστισμό τους ουσιαστικά σε τρίτες χώρες. Η εκπρόσωπος Ακνούρ μας είπε χθε ότι οι συμφωνίες αυτές είναι παράνομες. Μας ντροπιάζει η αύξηση του προπολογισμού για να τις τη στρατικοποίηση του Αιγαίου Πελάγους και όχι για τη διάσωση και την ανθρωπιστική υποδοχή των προσφύγων. Ούτε έχουμε ελαστικότητα για να προσαρμοστούμε στις ε, κατεπίκουσες ανθρωπιστικές ανάγκες και να δείξουμε την ελληνική μας. Ας μην απορρίψουμε τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για ένα λεπτό και πάλι. Ευχαριστώ. Ψήφισα κατά τη έκθεση αυτή, διότι επιβεβαιώνει την ε, νεοφιλελεύθερη στροφή των προπολογισμών. Ε, από την χρηματοδότηση, όλο και μικρότερη, ε, έως την έλλειψη του δημοκρατικού έλεγχου ο ευρωπαϊκό προπολογισμό προσανατολίζεται στην ενίσχυση τη οικονομική διακυβέρνηση και των δομών τη, ε, στηρίζοντα με δημόσια κονδύλια ε, απελευθερώσει ε, ε, κλάδων και μείωση των εργατσιακών δικαιωμάτων. Το τραγικό είναι ότι τα ίδια ε, κονδύλια ενισχύουν ταυτόχρονα μηχανισμούς της αγοράς αντί να δημιουργούν ένα αυτόνομο πόλο κρατικών επενδύσεων. Ε, ο το κράτος ε, επιδοτεί έτσι τις ιδιωτικές επενδύσεις. Ε, ε, εμείς θέλουμε ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Θέλουμε η Ευρώπη να ενισχύσει τα κονδύλια υπέρ των δημοκρατικών αποφάσεων των κρατών τους, αντί να τα εκβιάζει τα κράτη. Θέλουμε τα κονδύλια για την έρευνα ανάπτυξη στη βιομηχανία και τη γεωργία να κατευθύνονται στις τοπικές κοινωνίες και όχι στις αγορές. Ευχαριστώ. Χάναντ. Πριν από 800 χρόνια ένας βασιλιάς και κάποιοι βαρόνοι συμφώνησαν με δισταγμούς για να δημιουργήσουν ένα κοινοβούλιο στο Westminster. Η βασική λειτουργία του ήταν όχι η εκπροσώπηση, αλλά ο έλεγχος της κυβέρνησης. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά ζητήματα. Όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα. Η συζητήση, η εκπροσώπηση ε, του εκλογικού τους, <laughs> των πολιτών κλπ. Ε, ο στόχος του κοινοβουλίου ήταν ο έλεγχος. Κοιτάξτε τη διαφορά αυτού με όλα τα άλλα εθνικά κοινοβούλια όταν μιλάμε για τους προπολογισμού Και κοιτάξτε και τι κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, ως ευρωβουλευτές ε, ζητούμε όλο και περισσότερους ευρωπαϊκούς πόρους αυξήσει τον προπολογισμό. Αυτό ε, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να κάνουν οι, τα εθνικά κοινοβούλια, δεν δημιουργήθηκαν γι' αυτό. Ε, έτσι όπως πάμε, ο προϋπερασμός δεν πρόκειται ποτέ να μικρύνει, πάντα θα μεγαλώνει. Μα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είναι σχετικά σαφές ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού του 2017 θέλουν να εξορθολογήσουν την κατανομή των πόρων και τον προϋπολογισμό. Κάτι που είναι θετικό εν ώψη του 2020. Έχουμε την ψηφιακή αγορά, το πρόγραμμα Ερασμοσύν, προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και χρειαζόμαστε νέα προγράμματα, κυρίως στήριξη επιχειρηματικότητας. Αυτό είναι σημαντική προτεραιότητα και του κοινοτικού προϋπολογισμού. Είναι επίσης σαφές ότι χρειάζονται επιπλέον πόροι για την Ελλάδα, 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάτι τέτοιο θα μας δώσει μια νέα όθηση για να καταπολεμήσουμε την αστάθεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στίβεν Βόλφ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χθε στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Βουλή, ο Μαρκάνη, ο, ο διοικητή τη Τράπεζα τη Μεγάλη Βρετανία, είπε ότι ε, αν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατρέξει κίνδυνο. Αγνώρισε όμω ε, τον κίνδυνο τη παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κίνδυνο τη ε, απουσίας οποιασδήποτε αλλαγή εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα συζητήσαμε τι κατευθυντήρε γραμμέ για τον προπολογισμό το 2017 και λέμε ότι ε, θα πρέπει να αποτρέψουμε την διόγκωση του κοινωτικού προπολογισμού. Θα πρέπει οι Βρετανοί να καταλάβουν ότι θα ψηφίσουν ναι στο δημοψήφισμα, θα ψηφίσουν ναι σε μια οργάνωση που τη διοικούν δημόσιοι υπάλληλοι, που βασικό του μέλημα είναι να αυξήσουν τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί ε, ταυτόχρονα εκπροσώπηση. Και πολλές χώρες, ε, ε, πολλές, ε, πολλά κράτη απομακρύνθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο γιατί δεν, δεν ήθελαν φορολογία χωρίς εκπροσώπηση. Εδώ όμως θα έχουμε αυξήσει του προπολογισμού χωρίς να έχουν κανένα λόγο και καμία βαρύτητα στην απόφαση αυτή οι ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Στάνισλα Πόλτσακ. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση αυτή του κυρίου Γκάιερ, γιατί είναι πολύ σημαντικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού. Δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσταθεροποιηθεί σε έναν επιπλέον τομέα, δηλαδή το δημοσιονομικό. Η προηγούμενη Προεδρία του Λουξεμβούργου μας έδειξε πώς μπορούμε να εκπονούμε και να καταρτίζουμε αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς και μάλιστα να τους εγκρίνουμε κιόλας. Ήταν από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας. Και Ολλανδική Προεδρία αλλά και η Σλοβακική που θα ακολουθήσει να καταφέρουν να διεκπαιρεώσουν αισίως τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό. Χρειαζόμαστε μια ελαστικότητα στον προϋπολογισμό γιατί αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρές προκλήσεις. Στρατηγικές επενδύσεις, προσφυγική κρίση, εντάσεις ε, στη γειτονία μας. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις τελευταία ναι. επεξήγηση ψήφου για την έκθεση Γκάιερ ήταν αυτή και περνάμε στην επόμενη έκθεση της κυρίας Χιούμπνερ με θέμα τη Διοργανική Συμφωνία για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας. Κυρία Μορβάη, ε, απήχα από την ψηφοφορία αυτή. Υπάρχουν κάποια θετικά πράγματα σε αυτήν την έκθεση ιδιαίτερα η επιβεβαίωση της αναλογικότητας και της επικουρικότητας ε, και του ρόλου τους, όπως επίσης και η επιβεβαίωση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων. Ε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπενθυμίζουμε στους πολίτες μας πάντα τι σημαίνει η αρχή της επικορικότητας. Σημαίνει ότι τα, τα κράτη διατηρούν τις ε, ε, αρμοδιότητές τους ε, και δεν τις εκχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες ορίζονται με νομικά διάβλητο τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διακόπτει ο πρόεδρο. Ποιο Πόσπι, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα την έκθεση αυτή, διότι γνωρίζω πως ε, η ποιότητα των ε, νομοθετικών ασκημένων είναι αμφισβητούμενη πολλές φορές. Εγώ πολύ συχνά στη χώρα μου, τη Τσεχική Δημοκρατία, βλέπω διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας οδηγίας. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μεταγράφονται με διαφορετικό τρόπο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συμφωνία για την ε, ποιότητα του, της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας. Δεν είναι μόνο τεχνικό το θέμα. Ε, πολλές φορές είναι και ουσιαστικό το Κοινοβούλιο και, άλλα, τα άλλα θεσμικά όργανα ε, υποβάλλουν και εγκρίνουν νόμους χαμηλή ποιότητα. Αυτό επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών μα και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χαίρομαι που ενισχύεται ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ποσπίσιλ. Ο Σβέν Σούλτσε, για ένα λεπτό επίση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υπερψήφισα την έκθεση της κυρίας Χιούμπνερ, αλλά με κάποιες επιφυλάξεις και δυσκολίες. Ο προσανατολισμός της είναι σωστός, αλλά θα προτιμούσα περισσότερη σαφήνεια ε, και περισσότερες διευκρινήσεις επιμέρους σημεία. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, θα προτιμούσα ένα δεσμευτικό κείμενο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και επίση στι διαπραγματεύσει Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μεγαλύτερη διαφάνεια. Αν είμαστε έντιμοι, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την καλή αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κάπως αλλοιώθηκε στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Ψήφισε υπέρ, όπως σας είπα, αλλά με επιφυλάξεις παρόλα αυτά. Ο κύριος Μαμίκινης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά θα πρέπει να βελτιώσουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει η νομοθεσία μας να είναι υψηλών προδιαγραφών γιατί ούτως ή άλλως επηρεάζει τη ζωή 500 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στην Ιφίλιο και επηρεάζει και πολλούς τομείς, τον πολιτισμό, την υγεία, την παιδεία. Η συγκεκριμένη έκθεση είναι σημαντική και θα πρέπει να λάβει υπόψη τις πολλές πτυχές που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρομεσαίες. Οπότε η βελτίωση της νομοθεσίας και η απλούστευση της νομοθεσίας είναι επιθυμητές προθέσεις. Πολλοί ε, κόσμοι δεν έχει ιδέα τι γίνεται στα κοινοτικά θεσμικά όργανα. Θα πρέπει να έρθουμε πιο κοντά στους ψηφοφόρους μας. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και πρεψήφισε την έκθεση Χιούμπνερ. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Μακοβέ για ένα λεπτό. Ε, ε, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ πλούσια νομοθεσία. Μερικές φορές υπερβολική και ασαφής κάθε κράτος έχει τις δικές του προτεραιότητες και τα δικά του ενδιαφέροντα. Και μερικές φορές ε, η νομοθεσία επιτείνει το γραφειοκρατικό άχθος. Και μερικές φορές γίνεται ένα συνοθήλευμα διαφορετικών πραγμάτων, ε, κάτι που την κάνει πιο ε, δυσνόητη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν υπάρχει αρκετή συνοχή. Θα πρέπει οι νομοθετικές διατάξεις να είναι σαφείς, ακριβείς και σύντομες πάνω απ' όλα. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να θεσπίζουμε νομοθεσία υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών και όχι για να προωθεί ο καθένας τις δικές του προτεραιότητες. Αυτό θα, το κοινό συμφέρον θα πρέπει να είναι ο κοινό παρανομαστή όλων των νομοθετικών διατάξεων. Γι' αυτό Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχουν διαβουλεύσει και μεταξύ του αλλά και με του Ευρωπαίου πολίτε, εξασφαλίζοντα διαφάνεια. Ευχαριστώ. Μάρκους Πίπερ για ένα λεπτό. τώρα άνοιξε το μικρόφωνο. Ωραία. Ευχαριστώ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση Χούμπνερ. Είναι κάτι το θετικό. Η μείωση της γραφειοκρατίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουμε και την αξιολόγηση αντικτύπου της Κομισιόν. Όμως να υπενθυμίσω την πρόταση της Κομισιόν. Η Κομισιόν ήθελε να αποφευχθεί αυτός ο κανονιστικός υπερθεματισμός των κρατών μελών, ήθελε ευθύνη των κρατών μελών, ήθελε μια ετήσια λίστα νομοθεσίας που αποσύρεται. Γιατί λοιπόν Συμβούλιο και ειδικά το Κοινοβούλιο τα εμπόδισαν όλα αυτά σε μια νιρβάνα του τριμερούς ε, διαλόγου. Κάπου εκεί πέρα εξαφανίστηκαν. Η Κομισιόν ε, τώρα από ό,τι φαίνεται παίζει τον ε, μπαμπούλα της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας και είναι κρίμα πραγματικά άξιζε περισσότερα αυτή η συμφωνία. Ευχαριστώ Μάρκ Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, οι δεύτερη εκλεγμένοι ο σοσιαλιστές είναι κατά της ε, έκθεσης αυτής, γιατί προβλέπει μόνο διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Διαβούλευση, απλώς διαβούλευση, ενώ είμαστε συνομοθέτης. Δεν είναι αρκετό λοιπόν για ένα τόσο θεμελιώδη ζήτημα. Εξάλλου, οι σοσιαλιστέ πιστεύουμε ότι το τμήμα εκείνο που περιλαμβάνει στη συμφωνία αποτελεί ένα κίνδυνο και κινδυνεύει να καταστρέψει του κανόνε κοινωνική προστασία, περιβαλλοντική προστασία και δημόσια υγεία. Γι' αυτό λοιπόν για μα είναι απαράδεκτη μια τέτοια θεσμική συμφωνία. Η Ευρώπη σήμερα ασθενεί. Χρειάζεται κοινωνική ολοκλήρωση, νόμους που οδηγούν σε περισσότερη κοινωνική εναρμόνιση και το κείμενο αυτό δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις θεμελιώδεις ανάγκες. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, Στίβεν Βόλφε. Ευχαριστώ, κύριε την Πρόεδρε. Καλύτερη νομοθεσία, καλύτερη ρύθμιση. Ναι, κανείς δεν είναι κατά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θέλει, χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία. 40 χρόνια ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει οδηγήσει το ΕΠ των χωρών μας στα χαμηλότερα δυνατόν επίπεδα. Φυσικά, να μην έχουμε χαμηλή παραγωγικότητα, να μην υπάρχει ανεργία, να μην είναι 13% η ανεργία και ούτε πάνω από 30% η ανεργία των νέων σήμερα στην Ευρώπη. Είμαστε σε μια ήπειρο που αργοπεθαίνει εξαιτία τη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αν δείτε λοιπόν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, πρέπει να δείτε πώ δημιουργήθηκε αυτή. Στις Ηνωμένε Πολιτείε έχετε τους γερουσιαστές, έχετε τους βουλευτές οι οποίοι εκπονούν την νομοθεσία. Εδώ, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι αξιωματούχοι που εκπονούν την νομοθεσία. Φυσικά και χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία, αλλά είναι σαν το πλοίο που βουλιάζει και ο καπετάνιος φωνάζει «τρυπήστε περισσότερο το πλοίο». Ευχαριστώ. Τελείωσαν η επεξηγήση ψήφου για τη διοργανική συμφωνία και περνάμε στο ψήφισμα για τη συμφωνία με την Φίλιπ Μόρις. Η Κριστίνα Μορβά για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αν δείτε αυτή την έκθεση, τον τίτλο δηλαδή, λέει για συμφωνία για προϊόντα καπνού σε παρένθεση συμφωνία PMI και νομίζει κανείς ότι PMI είναι κάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, καμιά γραφειοκρατία, ε, κάποια συντομογραφία. Αν διαβάσει μόνο κανείς την έκθεση, καταλαβαίνει ότι PMI σημαίνει Philip Morris International. Η τεράστια αυτή η επιχείρηση καπνού και γίνονται τέτοιες συμφωνίες και με άλλες επιχειρήσεις. Θα πρέπει νομίζω να, να το δείχνουν αυτό στις εξετάσεις για το απολυτήριο Λυκείου. Ε, συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, PMI και αν δεν το καταλαβαίνουν ε, τότε δεν είναι έτοιμοι να αποφτύσουν και να είναι Ευρωπαίοι πολίτες ε, για να μάθουν το τι σημαίνει διαφάνεια και διαφθορά κτλ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, ο κύριος Πόσπισιλ. Αφού μελέτησα όλα τα έγγραφα, αισθάνομαι ότι πρέπει να δείξω επιφυλακτική στάση απέναντι στο έγγραφο. τα έγγραφα που έχω δείχνουν ότι η προηγούμενη συμφωνία ε, ήταν διαφορετική ε, ή μάλλον σήμερα ψηφίσαμε την παράτασή της. Από τη μία είχαμε μία μείωση της, του λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Από την άλλη όμως υπήρξε μία αύξηση των λεγόμενων λευκών τσιγάρων. Δηλαδή, η παράνομη κυκλοφορία των προϊόντων καπνού δεν μειώθηκε στην πραγματικότητα. Θα πρέπει νομίζω λοιπόν να βρούμε μια πιο συστημική λύση από μεμονωμένες συμφωνίες με κάποιες ε, εταιρείε παραγωγούς. Για να μην καταστρέψουμε και την νόμιμη αγορά προϊόντων καπνού στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριος Μάμικινς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Στη χώρα μου, την Λετωνία, τα πλαστά προϊόντα καπνού αυξάνουν κάθε χρόνο το μερίδιο τους όμως η περιφέρεια μας ανήκει στις πιο φτωχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο κόσμος προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί όσο δεν έχουν δουλειά έτσι θα παραμείνει η κατάσταση είναι κρίμα το ότι η Κομισιόν χρειάστηκε τόσο καιρό για μια τεχνική αξιολόγηση. Μόλις Φεβρουάριο του 2016 δημοσιοποιήθηκε το έγγραφο το οποίο περιμέναμε από πέρσι το Μάιο. Πρόκειται για παράνομο εμπόριο αυτό των ε, τσιγάρων ε, και χρειαζόμαστε οδηγίες για να περιορίσουν τη δραστηριότητα αυτή. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, Κλάους Μπουχνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μέχρι τώρα υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ της Φίλιπ Μόρης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ πως οι συμφωνίες αυτές πρέπει να αποφεύγονται επί της αρχής. Πρώτον, γιατί δεν ε, Ισραήλ χρήματα, δεύτερον γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συμφωνεί με μεμονωμένες εταιρείε. Υποτίθεται ασχολείται με όλες τις εταιρείε. Η βιομηχανία του καπνού προσπαθεί να επηρεάσει την πολιτική. Το βλέπουμε αυτό με την διαδικασία επιδιαιτησίας ε, που στην οποία προσφεύγει αυτή η εταιρεία ακριβώς για να επηρεάσει τους πολιτικούς. Πρέπει λοιπόν κατεπηγόντως να τραβήξουμε μία γραμμή, γι' αυτό χαίρομαι για το πώς ψήφισε το Κοινοβούλιο και τερματίστηκε αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, η κυρία Μακοβάη για ένα λεπτό. Uh, το παράνομο εμπόριο ε, προϊόντων ε, καπνού δημιουργεί απώλειες περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά μας χάνουμε. Πέρα από το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού, με αυτά τα χρήματα χρηματοδοτείται η παράνομη η διεθνής εγκληματικότητα, η σωματεμπορία, ε, και διάφορες άλλες παράνομες δραστηριότητες. Λυπάμαι πραγματικά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάστηκε τόσο χρόνο για να μας εξηγήσει ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής της συμφωνίας που έχει υπογραφτεί με τη Φίλιπ Μόρις. Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Θέλω να υπάρχει διαφάνεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις κανονικά έπρεπε να τηρήσουν σιγή νυχθείως. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έπρεπε κανονικά να δουν αυτά τα έγγραφα δεν, μπόρε, δεν μπόρεσαν να τα δουν παρά μόνο μέσα σε, ένα, σε μια αίθουσα δίπλα, διπλοκλειδωμένη αφού υπέγραψαν ένα κάρο χαρτούρα. Δώδεκα χρόνια πέρασαν από την πρώτη συμφωνία και το παράνομο εμπόριο προϊόντων καπνού έχει μεγεθυνθεί. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι αυτές οι συμφωνίες, αλλά διαφάνεια. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε άρα με τις επεξηγήσεις ψήφου διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 η ώρα.